Okay. I think this time. Proszę Państwa. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Po długim weekendzie μετά από ένα παρατεταμένο Σαββατοκύριακο μπορούμε να ξεκινήσουμε τις εργασίες μας ε, και την ημερήσια διάταξή μας. Να σας υπενθυμίσω, να σας υπενθυμίσω ότι σήμερα προβλέπεται και πρωινή και απογευματινή συνεδρίαση. Και η επόμενη μας ε, συνεδρίαση είναι την Πέμπτη το πρωί. Για να δούμε την ημερήσια διάταξη. Υπάρχουν παρατηρήσεις? Από ό,τι βλέπω όχι, οπότε εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Ε, η σημερινή μας συνεδρίαση μεταδίδεται μέσω του διαδικτύου και έχουμε διερμήνια σε 20 γλώσσες με εξαίρεση τα εστονικά, τα μαλτέζικα και τα σλοβακικά. Με την ε, κανονική διαδικασία θα εγκρίνουμε και τα πρακτικά της συνεδρίας της 14 η ως 16 Απριλίου και να περάσουμε ε, στην κοινή συζήτηση των σημείων 4 και 5 που αφορούν ε, παρόμοιο θέμα και δύο διαφορετικές χώρες, την ε, Μολδαβία και τη Γεωργία. Πρόκειται για την εφαρμογή μηχανισμού διασφάλισης κατά της καταστρατήγησης ε, που προβλέπει την προσωρινή αναστολή των δοσμολογικών προτιμήσεων τη Συμφωνία Σύνδεση μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομική Ενέργεια και των κρατών μελών τη αφενό και τη Μολδαβία αφετέρου για την πρώτη περίπτωση και τη Γεωργία για τη δεύτερη. Συντάκτης τη γνωμοδότησης ε, για το τμήμα τη Μολδαβία είναι η κυρία Νταντσίλα. Η δεύτερη γνωμοδότηση αφορά τη γεωργία. Ίδιο θέμα. Και πάλι από την 1η Σεπτεμβρίου εφαρμόζεται προσωρινά, όπως και η προηγούμενη συμφωνία. Αρμόδιος συντάκτης γνωμοδότηση είναι ο κύριος Νέκοφ. είναι παρόντες. Ε, οι συντάκτες νομοδότης ελπίζω ναι. Αν δεν έχετε αντίρρηση, ήθελα να συζητήσουμε από κοινού τα σημεία 4 και 5. Και πριν τη συζήτηση, υπάρχει ένα πρόβλημα όμως με τη βουλγαρική μετάφραση. Δεν ακούμε καλά την βουλγαρική διερμηνία. Έχει. Ένα λεπτό να το ελέγξουμε και τεχνικά το θέμα. Είσαι okay? Εντάξει τώρα. Ναι, ναι. Μια χαρά. Ωραία, όπω είπα λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι, θα συζητήσουμε από κοινού τα σημεία 4 και 5 και πριν ε, την έναρξη τη συζήτηση θα ήθελα να ζητήσω από τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, τον κύριο Σποτ Χάρη ε, από τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου και τον εκπρόσωπο της Γενική Διεύθυνσης Γεωργία, του καλωσορίζω στη συνεδρίαση και θα ήθελα να μα κάνουν μια ενημέρωση. Οπότε δίνω πρώτα το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρώτα. Και αν θέλει κάποιος να προσθέσει κάτι εκτός από εσά, το αφήνω στη διακριτική σας ευχαίρεια. Παρακαλώ, σας ακούμε. Thank you, Mr. Chairman. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να μπορέσουμε να σας δώσουμε κάποιες εξηγήσεις για τις προτάσεις μας για τις δύο αυτές ρυθμίσεις για την Γεωργία, τη Μολδαβία και τις ρήτρε προστασίας με τη Μολδαβία. Προέρχομαι από τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου Έχω και συναδέλφους από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και γι' αυτό αν έχετε ερωτήσεις αργότερα ίσως να μπορούμε να απαντήσουμε. Προτείνουμε δύο κανονισμούς λοιπόν σχετικούς με τη συμφωνία με τη Μολδαβία και τη Γεωργία. Οι κανονισμοί αυτοί στην ουσία θέτουν στο κοινοτικό δίκαιο κάποιες αποφάσεις των εταιρικών συμφωνιών με τις χώρες αυτές να σας εξηγήσω λίγο το γενικότερο πλαίσιο. Ορισμένες FTAs, τέτοιου είδους δηλαδή συνολικές συμφωνίες, περιλαμβάνουν ρήτρες και ειδικού μηχανισμούς. Απαιτείται λοιπόν μία νομική ρύθμιση έτσι ώστε οι μηχανισμοί αυτοί να τεθούν σε εφαρμογή λεπτομερώς. Ένα παράδειγμα. Διευκρινίζουν τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες οι μηχανισμοί οι ρήτρες προστασίας τίθενται σε λειτουργία. Διευκρινίζουν τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθηθούν και τη διαδικασία λήψεως αποφάσεων για τέτοιου είδους ρυθμίσεις. Όπως γνωρίζετε η συμφωνία με τη Μολδαβία εμπεριέχει και μια διμερή ρήτρα προστασίας και οι δύο επίσης συμφωνίες και με τη Μολδαβία και τη Γεωργία προβλέπουν έναν μηχανισμό για ορισμένα επεξεργασμένα γεωργικά προϊόντα. Οι προτάσεις για τους δύο αυτούς κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου έχουν κατατεθεί λίγο πριν τη σημερινή συνεδρίαση και αποτελούν την προτινόμενη νομική βάση, νομικό πλαίσιο μάλλον, για την εφαρμογή των δύο αυτών συστημάτων. Οι προτάσεις αυτές βασίζονται σε συγκρίσιμες ε, αντίστοιχες ε, ρυθμίσεις διακανονιστικές οι οποίες έχουν συμφωνηθεί στο παρελθόν για τις πρόσφατες εταιρικές συμφωνίες που είναι πλέον σε ισχύ. Παράδειγμα, βασίζονται στον κανονισμό για την Κορέα μετά από το FTA, την εταιρική συμφωνία με την Κορέα που έγινε δεκτή το 2011 την αντίστοιχη συμφωνία επίσης με την Κεντρική Αμερική, η οποία τέθηκε σε λειτουργία το 2013, όπως επίσης και τις συμφωνίες Κολομβίας και Περού για τις εταιρικέ συμφωνίες με τις δύο αυτές χώρες οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ το 2013. Καλύπτονται λοιπόν τα μέσα αυτά από τις νομικές ρυθμίσεις που ε, προτείνουμε. Όπως σας είπα, Πρώτον έχουμε ε, την διμερή ρήτρα προστασίας όπως ονομάζουμε. Το μέσο αυτό περιλαμβάνεται στη συμφωνία με τη Μολδαβία μόνον. Δεν υπάρχει αντίστοιχη τέτοια ρήτρα για τη συμφωνία με την Γεωργία. Ο λόγος είναι γιατί δεν υπήρξε διαπραγμάτευση στα πλαίσια της εταιρικής σχέσης με την Γεωργία για μια διμερή ρήτρα προστασίας στα πλαίσια της απελευθέρωσης εμπορίου ε, μια μεγάλη αύξηση των εισαγωγών μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σε αντίστοιχες οικονομικές δραστηριότητες ενός από τα δύο μέλη. Εφόσον δημιουργηθεί ένας τέτοιος κίνδυνος, τότε η διμερής ρήτρα προστασίας δίδει τη δυνατότητα είτε να αποκατασταθεί η προηγούμενη ε, ρύθμιση για τις δασμολογικές επιβαρύνσεις είτε να ακυρωθεί η αδίποτε περαιτέρω ε, φιλελευθεροποίηση της αγοράς στο συγκεκριμένα προϊόντα. Είναι αν θέλετε το τελικό δίκτυ προστασίας στην περίπτωση κατά την οποία η κατάργηση των δασμών οδηγήσουν σε σοβαρές βλάβες μέσω της ε, πολύ μεγάλης αύξησης των εισαγωγών. Η αύξηση των εισαγωγών είναι μια φυσιολογική συνέπεια βέβαια της φιλελευθεροποίησης του εμπορίου. Είναι ένα μέσο το οποίο τώρα πλέον είναι διαθέσιμο μόνο στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει ανεξέλεγκτη αύξηση των εισαγωγών. Κάτι το οποίο θα μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρή βλάβη στους παραγωγούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίδει την δυνατότητα στην οικονομική αυτή δραστηριότητα και στους γεωργούς ε, να αντιδράσουν, να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες, στις νέες καταστάσεις λόγω ακριβώς της απελευθέρωσης του εμπορίου. Πρόκειται δηλαδή το μέτρο το οποίο εμείς προτείνουμε για ένα προσωρινό ανακουφιστικό μέτρο που δίδει χρόνο στους παραγωγούς να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες εφόσον κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο. Ε, οι βασικές αρχές του συγκεκριμένου μέσου ανταποκρίνονται στις αντίστοιχες αρχές τις οποίες επιβάλλει ο ΠΟΕ. Δηλαδή λέγεται ότι εφόσον υπάρξει μια αυξημένη ε, ε, εισαγωγική, παρατηρήσουμε αυξημένες εισαγωγές, αυτές οι εισαγωγές θα μπορούσαν να δημιουργήσουν βλάβη στις τοπικές παραγωγές, στις εθνικές παραγωγές. Και φυσικά βέβαια αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να αποδειχθεί και να τεκμηριωθεί πριν ληφθεί το μέτρο. Τώρα για το πώς θα εφαρμοστεί η διαδικασία, εδώ κάποιες λεπτομέρειες. Υπάρχει καταρχάς μια διερευνητική περίοδος, η οποία ε, έχει διάρκεια εξαμήνου. Υπάρχει δυνατότητα στον κανονισμό παράτασης της ε, διερευνητικής αυτής περίοδου με ένα επιπλέον τρίμηνο, συνολικά εννέα μήνες, ανάλογα με την ε, περιπλοκότητα της έρευνας. Ε, υπάρχει επίσης η δυνατότητα επιβολής προσωρινών μέτρων τα οποία μπορεί να ληφθούν άμεσα, ε, να αποφασιστούν άμεσα ή και να ισχύσουν για μία μέγιστη περίοδο 200 ημερών. Είναι ένα πρώτο μέσο για την ε, ε, ανακούφιση, θα έλεγα, των παραγωγών σε περίπτωση που δημιουργηθεί μία απρόβλεπτη κατάσταση μέσω των αυξημένων εισαγωγών. <clears throat> Τα μέτρα αυτά λοιπόν μπορεί εφόσον αποφασιστούν με την κανονική διαδικασία να κρατήσουν δύο χρόνια. Εφόσον υπάρχουν συγκεκριμένες ε, προϋποθέσεις ε, υπάρχει δυνατότητα παράτασης της εφαρμογής τους για δύο ακόμα χρόνια, δηλαδή συνολικά τέσσερα. Αυτά τώρα να σας δώσω κάποιες ε, πληροφορίες για τον μηχανισμό αντικαταστρατήγησης. Αυτός ο μηχανισμός περιλαμβάνεται και στις δύο συμφωνίες, και για τη Μολδαβία και για τη Γεωργία. Οι προβλέψεις αντικαταστρατήγησης. Καλύπτει η πρόβλεψη αυτή τα γεωργικά προϊόντα. Στην περίπτωση κατά την οποία φτάσουμε ένα επίπεδο ανώτατο εισαγωγών για τα προϊόντα τα οποία περιλαμβάνονται στην συμφωνία, τότε οι δασμολογικές προτιμήσεις μπορεί προσωρινά να αναβληθούν για μία μέγιστη περίοδο 6 μηνών. Η αναβολή εφαρμογής, η διακοπή εφαρμογής θα ισχύσει στην περίπτωση κατά την οποία τα Υπουργεία Εμπορίου ε, δεν μπορούν να αποδείξουν ότι ε, τα προϊόντα αυτά είναι σαφές ότι προέρχονται από τα εδάφη τους. Οι ρυθμίσεις αυτές έχουν τεθεί σε ισχύ για να αποφύγουμε ακριβώς την δυνατότητα αποφυγής εφαρμογής των ρυθμίσεων στις εισαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή να μην έρχονται στην Ένωση μέσω της Γεωργίας και μέσω της Μολδαβίας προϊόντα τα οποία δεν είναι μολδαβικά ή γεωργικά. Απλά προσπαθούν να υποφεληθούν από τις ισχύουσες εμπορικές ρυθμίσεις. Και για τις δύο αυτές προτάσεις, κύριε Πρόεδρε, θα υπάρχει μια ετήσια έκθεση η οποία θα υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για το τμήμα το εμπορικό της συμφωνίας όπως επίσης και θα γίνονται παρατηρήσεις για την σωστή ή μη εφαρμογή των κανονισμών αυτών. Σχετικά τώρα με τις διμερείς ρήτρες προστασίας θα πρέπει να σας ενημερώσω ότι σε αντίστοιχες άλλες συμφωνίες ε, μέχρι τώρα δεν έχουν χρησιμοποιηθεί. Ε, υπάρχουν όπως σας είπα σαν ένα απότατο μέσο προστασίας στην περίπτωση κατά την οποία κάτι δεν πάει καλά στα πλαίσια της εφαρμογής των ρυθμίσεων της εμπορικής συμφωνίας. Είναι η πρώτη φορά που εισάγουμε ένα τέτοιο μηχανισμό σε μια εταιρική συμφωνία και προσπάθησα να σας εξηγήσω, ελπίζω να σας ενημέρωσα σωστά γιατί ε, το κάνουμε. Δεν έχω κάτι να προσθέσω, σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Φαντάζομαι αν ανακύψουν ε, απορίες ή ερωτήσεις, ε, θα σας ξαναδώσουμε το λόγο για να απαντήσετε. Τώρα θα δώσω το λόγο στους συντάκτες της γνωμοδότησής μας. Πρώτα στην κυρία Νταντσίλα, που είναι συντάκτρια γνωμοδότησης για το θέμα της Μολδαβίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε χαιρόμαστε για την πρόταση αυτών των μέτρων και αντιλαμβανόμαστε την ε, συνήθη διαδικασία για την προστασία των Ευρωπαίων παραγωγών σε ορισμένες περιπτώσεις για να μην κατακλειστεί η ευρωπαϊκή αγορά από τέτοια προϊόντα. Και μάλιστα η Ρουμανία ήταν η πύλη εισόδου των μολδαδικών προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά. Αλλά μέχρι στιγμής προβλήματα δεν υπήρξαν. Και είμαι βεβαία ότι δεν θα χρειαστεί καν να εφαρμόσουμε τον μηχανισμό διασφάλισης κατά της, κατα, της καταστρατήγησης. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι είναι απαραίτητος ένας τέτοιος μηχανισμός ε, που θα ενεργοποιηθεί όταν παραστεί ανάγκη. Είναι χρήσιμος ένα τέτοιος μηχανισμός και στις δύο συμφωνίες με τη Μολδαβία και τη Γεωργία. Επίσης Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό και θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες από την ε, Γενική Διεύθυνση Γεωργίας. Για τα βιομηχανικά προϊόντα μερικές φορές είναι πιο εύκολη η χνηλασιμότητα από ό,τι για τα απορροκυπευτικά. Γιατί εκεί ο τόπος παραγωγής ε, μερικές φορές είναι δυσκολότερο να ανοιχνευτεί. Τι σκοπεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει για τα γεωργικά αυτά προϊόντα για να εξασφαλίζεται η, ο εντοπισμός προέλευσής τους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Τώρα για την αντίστοιχη συμφωνία με τη Γεωργία θα δώσω το λόγο στον κύριο Νέκοφ. Παρακαλώ. Νέκοφ. Като цяло доклада мога да кажа, че е είναι πολυτεχνική φύσης η έκθεση αυτή και η συμφωνία η Συμφωνία Σύνδεσης ε, εφαρμόστηκε στην, την 1η Σεπτεμβρίου, αλλά από την Αύγουστο 2014 είναι τροποποιημένο το γεωπολιτικό πλαίσιο για τους ε, γεωργούς ό,τι αφορά και θέματα εξαγωγών από τη Ρωσική Ομοσπονδία. Πρέπει λοιπόν να τα αποκριθούμε στις ε, υποχρεώσεις μας ε, και σε ό,τι αφορά τη γεωργία. Οι ανησυχίες των ε, γεωργών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Θα πρέπει να υπάρξει μια απάνταση. Και από την μία πλευρά θα πρέπει να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας έναντι των εταίρων μας, αλλά αφετέρου πρέπει να μην παραμελήσουμε και τα συμφέροντα των δικών μας γεωργών, οι οποίοι επίσης θα πρέπει να υποστηριχτούν. Χρειαζόμαστε πιο πολλά στατιστικά στοιχεία για τα προϊόντα τα οποία εισάγονται από τη Γεωργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά εκ παραλληλού θα πρέπει να παρακολουθούμε την προέλευση των προϊόντων αυτών. Αν ισχύσει τελικά η ρήτρα αυτή. Τα προϊόντα θα πρέπει να εισαγάγονται χωρίς τελωνιακούς δασμούς στην περίπτωση αυτή. Και υπολογίζουμε στην ετήσια έκθεση για την παρακολούθηση της κατάστασης. Ευχαριστώ. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε. Περνάμε στη συζήτηση. Ο κύριος Μπούντα ζήτησε πρώτος το λόγο. Παρακαλώ, κύριε Μπούντα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Φυσικά, και εγώ Καλώς ορίζω την Επιτροπή και χαίρομαι για την παρουσία της εδώ. Χαίρομαι ιδιαίτερως και για τον ανοιχτό χαρακτήρα που επέδειξε κατά την ε, υιοθέτηση των συμφωνιών αυτών για τους ε, γεωργούς στην Μολδαβία και στην ε, Γεωργία. Και όπως είπε και ένας προηγούμενος ομιλητής, μας απασχολεί ιδιαίτερα το πώς θα προστατεύσουμε και τους δικούς μας γεωργούς. Γι' αυτό λοιπόν είναι τόσο κατάλληλος αυτός ο μηχανισμός σε ό,τι αφορά τις ε, νομικές διατάξεις και την προστασία που προσφέρουν. Θα μπορούσαμε με τον τρόπο αυτό να κρατήσουμε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης τα προϊόντα που δεν προέρχονται από τη Γεωργία και τη Μολδαβία. Είναι πολύ δύσκολο όμως για τα μη μεταποιημένα προϊόντα να εντοπίσουμε την προέλευσή τους. Δεν θα ήθελα λοιπόν αυτό, αυτή η ρήτρα Δικαιή ασφαλεία να χρησιμοποιηθεί με επιζήμιο τρόπο, να υπάρξει κατάχρηση δηλαδή τη ρήτρα αυτή. Γι' αυτό λοιπόν η ανιχνευσιμότητα των προϊόντων θα πρέπει να διαμορφωθεί στο σωστό πλαίσιο. Είναι πολύ τεχνική φύση η έκθεση, σύμφωνη, αλλά πιστεύω ότι έχουμε ένα σημαντικό ρόλο να δραματίσουμε εδώ για να διασφαλίσουμε ότι το εργαλείο αυτό τελικά θα καταστεί χρήσιμο και ωφέλιμο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Σουλαζό. Oui, Ευχαριστώ. Η ιδέα των ελεύθερων συναλλαγών με τρίτες χώρες που έχουν πολύ φθηνό εργατικό δυναμικό και πολύ χαλαρέ περιβαλλοντικέ και κοινωνικέ διατάξει, είναι επιβλαβείς τέτοιες συμφωνίε για τους Ευρωπαίους παραγωγούς εξαιτία του αθέμητου ανταγωνισμού και των στρεβλώσεων που δημιουργούνται. Αντί λοιπόν να έχουμε ε, ένα περίπλοκο μηχανισμό διασφάλιση και χρονοβόρο, γιατί πρέπει να περιμένουμε ζημίε στην οικονομία ενός περισσότερων χωρών. Γιατί λοιπόν να μην θεσπίσουμε ποσοστώσει στι εισαγωγέ αυτών των χωρών Πιστεύω ότι η λύση των ποσοστώσεων ε, θα απαλλάξει από το κίνδυνο της, τους Ευρωπαίους γεωργούς, ακόμη και αν ο κίνδυνος μερικές φορές είναι μικρός, και θα ε, αποφύγουμε την καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες γεωργούς. Καλύτερα πρόληψη παρά θεραπεία. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο λογικό αυτό. Άλλωστε στις, ε, στα γαλακτοκομικά προϊόντα και στις αγωγές κρέατος, ε, στις ε, συναλλαγές με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτή τη λύση προτιμήσαμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο παρακείμενός σας τώρα, ο κύριος Φεράντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ρήτρα προστασίας είναι μια καλή ενδιαφέρουσα ιδέα, αλλά δεν θα μπορέσουμε να την εφαρμόσουμε στην περίπτωση της Μολδαβίας, γιατί υπάρχουν συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών με τη χώρα αυτή. Ε, ρήτρες προστασίας για την κινέζικη εισβολή προϊόντων, ναι, αυτό θα το συζητούσαμε, αλλά νομίζω ότι Σήμερα στην Ευρώπη γίνονται πολλές καταστρατηγήσεις των ρυθμίσεων και στη Γεωργία, όχι υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπέρ άλλων χωρών που εποφελούνται από την χαλαρότητα την οποία έχουμε επιδείξει. Νομίζω ότι θα πρέπει εμείς να επανεξετάσουμε την αντίληψη την οποία έχουμε για την διεύρυνση και τη συνεργασία με τις γειτονικές χώρες και να επανεξετάσουμε τις οικονομικές μας σχέσεις με τις χώρες αυτές. Ευχαριστώ κύριε Σάγκνιο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να μας ε, διασφαλίσει, να εξασφαλίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο εκπρόσωπό ότι η Μολδαβία και η Γεωργία θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν αυτό το καθεστώς, το προνομιακό για το εμπόριο, αλλά όχι προκειμένου μεγάλες ε, χώρες να εξαγάγουν προϊόντα προς τη Μολδαβία, η οποία με τη σειρά να τα εξαγάγει εκ νέου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό που με απασχολεί ιδιαίτερα είναι τα αυγά. Θα ξέρετε πιο πολύ από εσά ότι σε ό,τι αφορά την παραγωγή στην Ευρώπη των αυγών δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ε, οι κλοβοί. Ωστόσο αυτό χρησιμοποιείται και στη Μολδαβία και σε άλλες χώρες. Άρα Φοβάμαι ότι τα αυγά αυτά θα μπορούσαν έτσι να επισέλθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, τα αυγά αυτά μπορεί να έχουν παραχθεί από τρόφιμα, από ζωοτροφές με συγκεκριμένα συστατικά τα οποία δεν χρησιμοποιούμε στις ζωοτροφές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί λοιπόν κατηγορηματικά να μου πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι αυτό αποκλείεται ως ενδεχόμενο. Państwa, <clears throat> nie mamy więcej zgłoszeń. Αυτά. Δεν βλέπω να ζητά άλλος κανείς το λόγο. Ο, α, συγγνώμη, ο κύριος Γλέζος. Γλέζος, πάνε πόσοι Γλέζος. Ε, αγαπητέ Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, μου είναι δύσκολο να παρακολουθήσω τη συζήτηση στις συγκεκριμένες χώρες το τι συμβαίνει δηλαδή με τα αγροτικά προϊόντα Μορδαβίας και Γεωργίας. Όμως θέλω να σας ενημερώσω για το τι συμβαίνει με την Ελλάδα, με τη χώρα μου, για να καταλάβετε τι πρέπει να αποφύγουμε ή τι πρέπει να προσφύγουμε. Σε τι πρέπει να προσφύγουμε. Δηλαδή, το κρασί Μπορντό θεωρείται ένα από τα γαλλικά ποτά τα πιο εξαίσια. Και όμως η παραγωγή ίνου στην Σαντορίνη, στη Σαντορίνη της Ελλάδας στέλνουν σε δεξαμενές στην, στο Αλγέρι από το Αλγέρι έρχεται στη Γαλλία και το ο μούστος της Σαντορίνης παρουσιάζεται σαν ποτό μπορντό της Γαλλίας. Είναι ένα φαινόμενο πασίγνωστο. Όπως και ένα άλλο σε ορυκτά προϊόντα. Περίφημα μάρμαρα της Ιταλίας Σκαράρα έχουν βγει από, την, από τα λατομεία της Νάξου. Γίνεται μία, ένα, υπάρχει ένα κομπρεμί κατά κάποιο τρόπο, υπάρχει μια μαφία κατά κάποιο τρόπο ανάμεσα στους εμπόρους που παίρνουν προϊόντα από μια άλλη χώρα και τα προσφέρουν ως προϊόντα μιας άλλης χώρας. Αυτό πώς θα καταπολεμηθεί. Αυτό είναι το πρόβλημα που με απασχολεί στην Ελλάδα. Σας δίνω τα στοιχεία και περιμένω να δω την απάντηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο. Κάθε χώρα να είναι γνωστό γνωστά τα προϊόντα της και να μπορεί να μην τα εκμεταλλεύεται άλλη χώρα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ξέρετε, η παγκοσμιοποίηση, το άνοιγμα των αγορών ε, έχει αυτά τα επιζήμια αποτελέσματα που επισημάνατε κι εσείς τίποτα δεν υπάρχει πια Java δωρεάν, δεν προσφέρεται τίποτα. Θα ήθελα τώρα να ζητήσω από τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αν θέλει να απαντήσει και κατόπιν και στους δύο συντάκτες μας ίσως να δευτερολογήσουν. Ο, εκπρόσωπο εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρακαλώ. Um, thank you, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και για τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και κάποιες ερωτήσεις που θέσατε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλα τα σχόλια και ελπίζω να με βοηθήσουν και οι συνάδελφοι. Ένα από τα θέματα που ακούσαμε. Πώς καθορίζεται και πώς θα καθορίζεται η προέλευση των γεωργικών προϊόντων. Σωστά επισημάνθηκε ότι τα βιομηχανικά προϊόντα είναι πιο απλό και εύκολο να καθοριστεί η προέλευσή τους. Αλλά πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορέσει να παρακολουθήσει το θέμα της προέλευσης των γερικών προϊόντων. Είναι πολύ καλό το ερώτημα αυτό. Εύλογο. Αλλά για το λόγο αυτό ακριβώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις δύο συμφωνίες αυτές διαπραγματεύτηκε αυτό το μηχανισμό κατά της παρέμβασης, καταστρατήγησης. Αυτός ο μηχανισμός καταστρατήγησης έχει προγραμματιστεί για να ελέγχει τον όγκο εισαγωγών και να διασφαλίζει ότι οι εισαγωγέ αυτέ και ο όγκο των εισαγωγών συνάδουν με τον όγκο παραγωγή τη κάθε χώρα. Μέσω στατιστικών στοιχείων λοιπόν που θα έχει στη διάθεση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορέσει να παρακολουθεί, να υποπτεύει τους όγκους των διαφόρων προϊόντων, των γεωργικών και μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων που προέρχονται από τις δύο χώρες αυτές. Αν οι ποσότητες αυτές φαίνεται ότι υπερβαίνουν τα φυσιολογικά όρια και τους όρους και τους όγκους που προβλέπονται στη συμφωνία, έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη δυνατότητα να ζητήσει από τις ε, χώρες εξαγωγής να αποδείξουν την προέλευση των επιπρόσθετων ποσοτήτων που εισαγάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι σχεδιάστηκε ο μηχανισμός αυτός για να αποφύγουμε έλεγχο κάθε παρτίδας που θα ήταν και χρονοβόρο και θα σήμαινε πολύ μεγάλο κόστος. Άρα το σύστημα αυτό βασίζεται στον έλεγχο των ποσοτήτων που εισάγονται. Κάποιος άλλος μίλησε και για τη ρίστα προστασίας, τη διμερή ρήτρα προστασίας. και αναφέρθηκε και στο χρόνο αντίδρασης, ο οποίος ενδεχομένω δεν είναι υπερβολικά μεγάλος αυτό το διάστημα αντίδρασης. Να πω, στην παρούσα φάση, ότι η διαδικασία, όπως προβλέπεται στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προβλέπει και μία διαδικασία κατεπήγοντος. Μία διαδικασία με την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί τάχιστα να λάβει αποφάσεις σε περίπτωση ε, εξαιρετικών περιστατικών για να προστατεύσει τα συμφέροντα των καλλιεργητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ισχύει και για τον ε, μηχανισμό καταστρατήγησης. Αυτή η διαδικασία κατεπήγοντος. Κάποιος επίση αναφέρθηκε και στην ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπή Όντω, και οι δύο χώρες θα αποτελέσουν αντικείμενο λεπτομερέστατη ετήσια έκθεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα περιλαμβάνουν όλες τις πτυχές των ε, συμφωνιών αυτών σε βάθος θα υπάρχουν λεπτομέρειες για τα στατιστικά στοιχεία, για τις εξελίξεις των ροών, για τους ποσότητες εξαγωγών. Λεπτομερείς πληροφορίες επίσης σε περίπτωση που ο μηχανισμός καταστρατήγησης και ρήτρα προστασίας έχουν τεθεί σε εφαρμογή. Ευχαριστώ. Παρακαλώ και συνάδελφό σας. Συγγνώμη, ξεχάσαμε μία ερώτηση για τα παρακυβευτικά. Θα την απαντήσει ο συνάδελφος που είναι ειδικό στα γεωργικά προϊόντα. Ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η συγγήτρια από τη Μολδαβία ρώτησε για τα απορροκυπευτικά από τη Μολδαβία. Μιλάμε για δαμάσκηνα, σταφύλια και μήλα για να σας αναφέρω την χρήση για το 2014 για τα σαφίλια έχουμε 42% της ποσόστοσης για τα μήλα κάτω από 1% της χρήσης ε, ποσοστώσεων για τα δαμάσκηνα είχαμε 700 τόνους 7% μόνο της ποσόστοσης Ευχαριστώ Λίγο Thank Κύριε Πρόεδρε, έγινε κάποιες αναφορές για την παραγωγή. Να πω το εξή, ότι το 2009 μέχρι το 2012 η Μολδαβία δεν εξήγαγε, δεν εξήγαγε στην Ευρώπη. Στην υπόλοιπη Ευρώπη 207 τόνους στην στον υπόλοιπο κόσμο. Αυτά για τη Μολδαβία. Και αυτό και για τη Γεωργία. Δεν είναι σημαντικέ οι εξαγωγέ αυτέ. Κάτι αναφέρθηκε τώρα για τις πρωτεΐνες ε, σε ό,τι αφορά τα αυγά. τις πρωτεΐνες που χρησιμοποιούνται για τις ζωοτροφές. Σας ευχαριστώ κύριε Αγνιό. Ο... Έθεσε ένα θέμα νομίζω λέει ο πρόεδρος για τα αυγά στα μεταποιημένα προϊόντα. Όχι μόνο γενικά για τα αυγά που εισαγάγονται από τη Μολδαβία αλλά σε ό,τι αφορά τα μεταποιημένα προϊόντα. Τουλάχιστον εγώ αυτό κατάλαβα από την ερώτησή σας, κυρία Γνιό. Για να είμαι δίκαιος, δεν ήταν κακή η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά δεν έγινε διάκριση μεταξύ της πρώτης ύλη και των μεταποιημένων προϊόντων. Αν θα θέλετε λοιπόν να διευκρινίσετε και αυτό το ζήτημα. Ναι, το είπα και εγώ αυτό το επισήμενο. Ο κύριος Ντες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ζήτησα το λόγο. Γιατί δικαίω ε, αναφέρθηκε ότι θα πρέπει να ισχύουν οι ίδιοι όροι και οι ίδιε διατάξει από αυτέ που ισχύουν στην Ευρώπη. Να υπογραμμίσω παρά όλα αυτά ότι στην Ευρώπη χρειαστήκαμε πάνω από 40 χρόνια για να έχουμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση τις ίδιες και πριν από λίγα χρόνια μόλις καταφέραμε να περάσει νομοθεσία για τα φυτοπροστατευτικά. Πριν από τη φάση αυτή ήταν πολύ διαφορετική η όρη που ίσχυαν σε όλη την Ευρώπη. Θα πρέπει φυσικά να βρούμε σωστές λύσεις και οι χώρες αυτές θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να εισάγουν στην Ευρώπη. Μίλησα με τον ε, Μαροκινό Υπουργό Γεωργίας και ξέρω ότι μας δίνουν και μας εξάγουν ντομάτες οι Μαρόκοι και δεν ήταν τόσο ενθουσιασμένοι οι Γάλλοι, οι Ιταλοί, οι Ισπανοί. Αλλά μου είπε ο Μαροκινός υπουργό κάτι το οποίο με εντυπωσίασε. Μου είπε ότι είτε θα έχουμε τη δυνατότητα να σας δίνουμε προϊόντα ή θα έρθουν προς εσάς οι νέοι μας θα πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία στους ανθρώπους αυτούς να μπορέσουν να αναπτυχθούν μέσα του εμπορίου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προκειμένου να έχουν μια προοπτική και οι νέοι στις χώρες αυτές. Να υποστηρίξουμε λοιπόν μια ισορροπημένη συμφωνία η οποία να είναι αποδεκτή και από τις δύο πλευρές. Τα σχόλιά σας κύριε δείχνουν ότι για πολλά θέματα της κοινή γεωργικής πολιτικής ε, ότι πολλά θέματα μάλλον της πολιτικής, της κοινή πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτώνται από εξωτερικούς παράγοντες. Αλλά είπαμε, παγκοσμιοποίηση. Είναι λογικό να υπάρχουν αλληλεπιδράσεις και να επηρεαζόμαστε και από τις εξωτερικές συνθήκες. Η κυρία Νταντσίλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις πληροφορίες και τις απαντήσεις τις οποίες έδωσε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για την δική τους συμμετοχή και συνεισφορά. Συμπερασματικά αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι οι συγκεκριμένες αυτές ρυθμίσεις απαιτούνται θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, το γεωπολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούμεθα. Τα μέτρα αυτά τα οποία θα θέλαμε να μπορούμε να εφαρμόζουμε θα πρέπει να είναι στη διάθεσή μας, θα πρέπει να υπάρχουν και η ρήτρα προστασίας και ο μηχανισμός αντικαταστρατήγησης για να μην υπάρχει έστω και μία αμφιβολία σχετικά με την επιθυμία προστασίας των Ευρωπαίων παραγωγών. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, περιμένω και γραπτές προτάσεις αν έχετε. Ε, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σνέκοφ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ακούσαμε αρκετές ενδιαφέρουσες απόψεις. Ο κύριος Ντες είπε ότι θα πρέπει να επιλέξουμε ανάμεσα στις ντομάτες από τη μία και τους πρόσφυγες από την άλλη. Θα πρέπει κυρίως όμως να προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε ε, τους ε, ε, παραγωγούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους γεωργούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή πρέπει να είναι η προτεραιότητά μας και γι' αυτό ακριβώς απαιτούνται αυτού του είδους οι ρήτρε προστασίας, έτσι ώστε να υπάρχει ε, μια ισορροπημένη ανάπτυξη όχι μόνο των σχέσεών μας με τις γειτονικές χώρες, αλλά στο ίδιο το εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοιτάξτε, οι δύο αυτές ρυθμίσεις εκθέσεις είναι τεχνικής φύσεως. Ε, κάποιες επιμέρους λεπτομέρειες παραμένουν σε εκκρεμότητα. Ελπίζω ότι σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταλήξουμε σε μία κάποια λύση. Ε, η προτεραιότητά μας είναι η προστασία των ευρωπαϊκών προϊόντων και γι' αυτό ακριβώς έχουμε κάνει και αυτές τις ρυθμίσεις για τη Μολδαβία και τη Γεωργία. Ο κύριος Ντέσσα θα προσθέσει μία ακόμη φράση. Επειδή αναφέρθηκε το επιχείρημά μου, θα ήθελα με την παρέμβασή μου ε, να πω ότι σε καμία περίπτωση δεν υπονομεύω την προστασία του καταναλωτή. Είναι ύψη τη σημασία και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ασφαλώ. Απλά μία διευκρίνηση να κάνω αυτό. Σα ευχαριστούμε. Οπότε ολοκληρώνουμε τη συζήτηση των δύο αυτών σημείων, 4 και 5. Το χρονοδιάγραμμα σας έχει διανεμηθεί. Και μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο, δηλαδή το 6, που προβλέπει ανταλλαγή απόψεων με εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ρωσικό εμπάργο και τις συνέπειες του στην αγορά οποροκυπευτικών. με πρωτοβουλία του συναδέλφου Ραμόν Λουίς Βαλκάρσελ Σίσο, που είναι αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Καταλήξαμε στην ανάγκη να ζητήσουμε πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα του ρωσικού εμπάργου και των συνεπειών του στην αγορά φρούτων και λαχανικών για τους Ευρωπαίους παραγωγούς που υπέστησαν πολλές ζημιές. Πολλά και ασχοληθήκαμε με το θέμα του ρωσικού εμπάργου περισσότερο για τα γαλακτοκομικά στις χώρες της Βαλτικής ε, ή τα φρούτα της Πολωνίας, αλλά έχουμε κοινή αγορά. Δεν είναι μόνο αυτές οι χώρες που επηρεάζονται από το ρωσικό εμπάργο και άλλες χώρες επηρεάζονται από το ρωσικό εμπάργο, κυρίως οι χώρες του Νότου, που έχουν άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Οπότε θα πρέπει να δούμε τα προβλήματα υπό το πρίσμα διαφορετικών ευρωπαϊκών περιφερειών, γιατί κάθε περιφέρεια έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και τις δικές της παραγωγές. Γι' αυτό και παρακαλέσαμε και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και δύο εκπροσώπους από τον τομέα οποροκυπευτικών από την περιφέρεια της Μούρσιας στην Ισπανία, ε, να μας παρουσιάσουν την κατάσταση. Πρώτα θα δώσω το λόγο στον ε, κύριο Παρκαβέλα. Ο κύριο Βαλκάρσης ο δυστυχώ δεν έχει έρθει ε, λόγω των ε, περιφερειακών και τοπικών εκλογών που έγιναν ε, προχθέ στην Ισπανία. Είχαμε και εμεί στην Πολωνία δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών. Εξελέγει ο κύριο Ντούντα, ευρωβουλευτή από την ομάδα των μεταρρυθμιστών και συντηρητικών. Αλλά μην ξεχνάμε ότι έχει μεσολαβήσει και ένα χρόνο από τις ε, δικέ μα εκλογέ ευρωεκλογέ. Έχει ήδη περάσει σχεδόν ένας χρόνος. Θα ήθελα να δώσω το λόγο πρώτα στον Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Άγκρη, τον κύριο Γιάννη Σχάπς, που θα μας ενημερώσει και κατόπιν εκπροσώπους το τομέα απορροκυπευτικών από τη Μούρσια. Uh, ευχαριστώ, Και συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια και για τα αποτελέσματα στην ε, Πολωνία. Πιστεύω ότι είναι απόλυτη αναγκαιότητα να συζητήσουμε τα αποτελέσματα των διαφόρων μέτρων σε ό,τι αφορά την απαγόρευση της Ρωσικής Ομοσπονδίας από 1η Αυγούστου του 2014. Γνωρίζουμε επίσης ότι αυτό δεν αποτέλεσε μόνο πρόβλημα για τα οποροκυπευτικά, αλλά και για άλλους τομείς οι οποίοι επηρεάστηκαν σημαντικά σε ό,τι αφορά τα γαλοκτομικά, τα πουλερικά, τα αυγά και πολλά άλλους τομείς. Και νομίζω ότι αυτό αποτέλεσε μία από τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε ως θεσμικά όργανα. Το πώς θα βοηθήσουμε τους παραγωγούς να προσαρμοστούν στη νέα κατάσταση. Η οποία σίγουρα επηρεάστηκε από το περιφερειακό πλαίσιο και από τα διάφορα προϊόντα, τα ανεκταρίνη, τα μήλα και πολλά άλλα και τη διάφορο, τα διάφορα μερίδια, αν θέλετε, ανακράτως μέλος σε ό,τι αφορά τα προϊόντα τα ρωσίκα όπου είχαμε ουσιαστικά 100% απαγόρευση. Νομίζω ότι καταφέραμε σχετικά γρήγορα να πάρουμε μέτρα κατεπήγοντος χαρακτήρα, εξαιρετικά μέτρα, με άμεση θέση σε ίσχυ, με πράξη κατεξουσιοδότηση, με απότερο σκοπό να σταθεροποιήσουμε την δύσκολη κατάσταση στην αγορά προτείναμε συγκεκριμένα μέτρα τα οποία στη συνέχεια εφαρμόστηκαν στο επίπεδο κράτων μελών σε ό,τι αφορά απόσυρση από την αγορά, προώθηση. Έγινε επίσης απόσυρση και για ελεύθερη διανομή. Μέτρα μη ε, συγκομιδής ή πράσινης συγκομιδής σε ό,τι αφορά λοιπόν την ε, εισαγωγή στην αγορά. Τα πρώτα μέτρα εφαρμόστηκαν ε, αρκετά γρήγορα το καλοκαίρι ήδη. σε ό,τι αφορά την συνέχεια της συγκομιδής το 2014 και τώρα κοιτώντας τα συνολικά στοιχεία, διαπιστώνουμε ότι περίπου 700.000 τόνοι τροφίμων αφαιρέθηκαν από την αγορά και μιλάμε για 120 έως 150 εκατομμύρια ευρώ βοήθεια που δόθηκε στους ε, παραγωγούς και στους ε, αγρότες. Θα ήθελα να πω ότι από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθήσαμε τάχιστα να βρούμε άλλους προορισμούς στον κόσμο. Ξέρουμε ότι η Ρωσία αποτελούσε πολύ σημαντικό προορισμό για εξαγωγές από τρετές χώρες, όχι μόνο για απορριπευτικά, αλλά και για προϊόντα γαλακτοκομικά και κρέατος. Και νομίζω ότι συνολικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατάφερε με επιτυχία να ανοίξει νέες αγορές η Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΤΕ που είναι αρμοδία για θέματα φυτοπροστασίας και οι συνάδελφοι στη Γενική Διεύθυνση Trade Εμπορίου με τις πρωτοβουλίες πρόσβασης στην αγορά μας ε, βοήθησαν στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας για να πετύχουμε εξαγωγές τις οποίες δεν είχαμε στο παρελθόν υπό κανονικές συνθήκες. Για κάποια προϊόντα, όπως για παράδειγμα στα μήλα, η Βραζιλία, η ΙΠΑ, ακόμα και η Μέσα Ανατολή Καταφέραμε λοιπόν να αποστείλουμε πολύ πιο μεγάλε ποσότητε από τις ε, κανονικέ. Σε ό,τι αφορά τις τιμέ, δε, ναι, οι τιμέ ήταν πιο χαμηλέ από ότι τα προηγούμενα χρόνια, ιδιαίτερα για τα μήλα, αλλά με μία μικρή διαφορά και για τι ντομάτε και για τα αχλάδια και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη σε κάθε περίπτωση ότι το 2014 ήταν ένα ιδιαίτερο έτος σε πολλές ε, περιοχές. Είχαμε καρπούς ε, της Πάμπας. Υπάρχει και το θέμα της παραγωγής ε, και συγκομιδής αχλαδιών και μήλων και είχαμε 10% παραπάνω παραγωγή από τα προηγούμενα έτη. Αυτό ασφαλώς αποτέλεσε μια επιπρόσθετη περιπλοκή και πρόκληση. προκειμένου να βρεθούν τα σωστά μέτρα για να υπάρχουν να υπάρξει διοχέτευση σε άλλες αγορές παρά το γεγονός ότι ο βασικός προορισμός κατά το παρελθόν ήταν η Ρωσία. Για κάποιες χώρες πιο σημαντικός προορισμός και από ότι η εσωτερική αγορά. Ξέρουμε επίση ότι και η ιστορική κατανάλωση θα μπορούσε να είναι καλύτερη. Ξέρουμε από τα στατιστικά στοιχεία ότι η παραγωγή οπροκυπευτικών μειώνεται συνολικά. Και καταβάλαμε σημαντική προσπάθεια να προωθήσουμε την κατανάλωση μήλων. Είδατε εκστρατείε, ιδιαίτερα και στο Βέλγιο. Έχουμε διάφορες εκστρατείε που θα μπορούσαμε να προωθήσουμε σε συνάρτηση και με τις ιδιαίτερες συνθήκες που σημειώθηκαν την περσινή χρονιά για να υπάρξει περαιτέρω κατανάλωση που δεν θα υπήρχε σε κάθε περίπτωση ενδεχομένω αν δεν υπήρχε η απαγόρευση εξαγωγής προς τη Ρωσία. Να υπογραμμίσω επίσης ότι το εμπόριο είναι καινοτομικό. Σίγουρα θα έχετε δει κάποια αριθμητικά στοιχεία που προκαλούν έκπληξη. Για παράδειγμα, εξαγωγές στη Λευκορωσία, οι οποίες αυξήθηκαν ραγδαία. Πιστεύουμε ότι ακόμα και αν τα στοιχεία άμεσου εμπορίου με τη Ρωσία πήγαν από το 95-99%. Μπορεί να πετύχαμε επιπρόσθετες ποσότητες με άλλες αγορές πέρα της Ρωσικής. Μέσω των εξαγωγών σε γειτονικέ χώρες. Τι εξαγωγούμε συμπέρασμα λοιπόν από την πρωτοβουλία αυτή έως τώρα. Με ένα συνδυασμό διάφορων μέτρων θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να πετύχουμε σταθεροποίηση της κατάστασης τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο τους τελευταίους εννέα μήνες. Δεν ε, ισχυρίζομαι ότι καταφέραμε να το κάνουμε αυτό κατά τη διάρκεια της συγκομιδής. Ιδιαιτέρως στην Κεντρική Ευρώπη ήταν δύσκολη κατάσταση για φαμίλα και επίσης αντιμετωπίσαμε δυσκολίες εφαρμογής κάποιων μέτρων όπως θεωρούσαμε ότι θα έπρεπε να εφαρμοστούν. Είμαι όμως αρκετά αισιόδοξο. Πιστεύω ότι τα προβλήματα αυτά επιδιορθώθηκαν τους πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους. Και κοιτώντα τώρα τις τιμές των μήλων, για παράδειγμα, στην Πολωνία, πιστεύω ότι η κατάσταση είναι αρκετά καθυσυχαστική. Το επίπεδο των τιμών είναι αρκετά υψηλό ίσως και υψηλότερο από το επίπεδο των τιμών την περσινή χρονιά. Ένα δεύτερο στοιχείο, επίσης σημαντικό, είναι ότι οι, οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βρήκαν άλλες αγορές εξαγωγής. Ήταν κάτι καινούριο αυτό το στοιχείο. Γιατί ξαφνικά διαπιστώσαμε την ανάγκη και για τα θεσμικά μας όργανα να είμαστε πιο ενεργοί, να ανοίξουμε για αγορές που έμειναν κλειστές ιδιαίτερος ε, λόγω των ε, φυτοπροστατευτικών μέτρων. Σε κάποιες περιπτώσεις σημειώσαμε επιτυχία, αφαιρώντας τέτοια μέτρα φυτοπροστατευσίας, αλλά σε άλλες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα η συμφωνία με την ε, Κορέα για τα ζωικά προϊόντα, εδώ πέρα δεν μιλάμε τόσο πολύ για προκυπαστικά, αλλά και η Βραζιλία αποτελεί νομίζω καλό παράδειγμα οι Βραζιλιάνοι δεν ε, αγόραζαν μήλα. Εδώ λοιπόν πιστεύω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να εξετάζουμε τι άλλες δυνατότητε υπάρχουν. Και θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη σε κάθε περίπτωση το γεγονός ότι το ευρώ και η αναλογία με το ισοτιμία με, την, με το δολάριο δυσκόλεψε περαιτέρω τα πράγματα. Αλλά μας επέτρεψε να εξαγάγουμε με ανταγωνιστικές τιμές στα προϊόντα μας. Είχαμε πραγματικά συγκομιδή ρεκόρ το 2014. Ιδιαίτερα για τα μήλα. Για τη φετινή χρονιά τώρα, μια μικρή πρόβλεψη, γνωρίζοντας τον κλάδο Σίγουρα λόγω της ε, παραγωγής ε, και λόγω της εναλλαγής των ετών παραγωγής και συγκομιδής θα είναι πιο χαμηλή η παραγωγή. Ένα δεύτερο στοιχείο που είδαμε, τα αριθμητικά στοιχεία για τα νεκταρίνια και για τα ροδάκινα, είναι πολύ μικρές οι διαφορές σε σχέση με την περσινή χρονιά, Άρα δεν αναμένουμε στο σημείο αυτό ουσιαστικές αλλαγές στα επίπεδα παραγωγής. Αλλά όπως ξέρετε όλα αυτά εξαρτούνται και από τις καιρικέ συνθήκες. Ελπίζουμε λοιπόν να έχουμε καλή σόδια για τους ε, αγρότες μας. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Αλλά Συχνά οι γεωργοί λένε ότι όσο καλύτερε είναι οι εισοδιέ, τόσο μεγαλύτερη είναι η κρίση μερικές φορές. Τώρα θα δώσω το λόγο στους εκπροσώπους των οργανώσεων ε, παραγωγών απορροκυπευτικών της Ισπανίας, της Μούρσια. Η κυρία Έστερ Γκόμες θα πάρει πρώτα το λόγο, που είναι αντιπρόεδρος ε, της οργάνωσης. Παρακαλώ μην ξεπεράσετε το πεντάλεπτο στις παρουσιάσεις σας για να έχουμε αρκετό χρόνο για, τις, ε, για τη συζήτηση, τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις. Γιατί δεν έχουμε περιόριστο χρόνο για το σημείο αυτό. Μάλιστα το υλικό που ετοιμάσατε για την παρουσίαση μπορούμε να το μοιράσουμε σε ευρωβουλευτές. Γιατί βλέπω πολύ ενδιαφέρον υλικό και πλούσιο. Αλλά παρακαλώ να είστε πολύ πιο σύντομοι στην παρουσίασή σας. Μία σύνοψη να μας κάνετε. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω θερμά την Επιτροπή σας για την ευκαιρία που μας δίνετε να λάβουμε το λόγο και να σας παρουσιάσουμε το σοβαρότατο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Θα ήθελα να σας πω ότι εγώ εκπροσωπώ και θα σας παρουσιάσω τις απόψεις όλων των Ισπανών παραγωγών, αλλά και των Γάλλων και Ιταλών που έχουν παρόμοια προβλήματα. Και την τελευταία χρονιά πολλές φορές είχαμε συνομιλίες με Ιταλούς και Γάλλους συναδέλφους προκειμένου να αναλύσουμε την κατάσταση και να κάνουμε διάγνωση αυτής. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω κύριε Πρόεδρε ότι σε σχέση με αυτά που μας είπε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ήθελα να διευκρινίσουμε ότι στα φρούτα με πυρήνα, με καρπό, δεν υπήρξε αρκετός χρόνος για το άνοιγμα των αγορών, γιατί μέσα σε ένα χρόνο είναι σχεδόν αδύνατο να επιστρέψουμε στην προηγούμενη κατάσταση. Όπως είπαμε και είδαμε και χθε, η κατανάλωση αυτών ε, των πυρηνόκαρπων ε, έχει αποτελματωθεί και οι τάσεις ε, των τιμών είναι χαμηλές γιατί υπάρχει υπερβολική προσφορά. Τα γεωργικά εισοδήματα των περισσότερων παραγωγών προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά από τις πωλήσει των γεωργικών τους προϊόντων. Στην περίπτωση των Ισπανών, για παράδειγμα, τα φρούτα αποκλείστηκαν από το καθεστώς ε, ενιαίας ενίσχυσης. Οπότε έχουμε πολλούς φραγμούς στην προσπάθεια αναζήτησης τρίτων αγορών. Στην περίπτωση των εξαγωγών, των ισπανικών εξαγωγών, Συγγνώμη, έχουμε ένα πρόβλημα με τις διαφάνειες εδώ. Λυπάμαι. Λοιπόν, οι ισπανικές εξαγωγές φρούτων και λαχανικών στις υπόλοιπες ε, χώρες δεν έχουν απορροφηθεί. Ε, δεν έχουν ε, αντικαταστήσει οι εξαγωγές προς τρίτες χώρες τις εξαγωγές που χάσαμε προς τη Ρωσία. Οι προβλέψεις των τιμών για το 2015 είναι ίδιες με αυτές του 2014 και συγκεκριμένα. Θα ήθελα να τονίσω ότι ήταν κατακόρυφη η πτώση ε, των ε, δαμάσκινων, ε, ροδάκινων και νεκταρινιών. Οπότε θα πρέπει κατεπηγόντως να ληφθούν μέτρα για τα προϊόντα αυτά. Γιατί οι παραγωγοί δεν μπορούν να αντέξουν αυτή την κατάσταση, την οποία δεν προκάλεσαν οι ίδιοι και είναι απλώς τα θύματα της. Σε ό,τι αφορά το άνοιγμα των αγορών, επαναλαμβάνω, είναι σχεδόν αδύνατο να απορροφηθούν οι εξαγωγές ε, που είχαμε προς τη Ρωσία. Θα πρέπει να εφαρμόσουμε την αντίστροφη στρατηγική. Δηλαδή, ό,τι ό,τι απαγορεύεται δεν επιτρέπεται μάλλον ό,τι δεν απαγορεύεται επιτρέπεται, εννοεί η ομιλήτρια, και έτσι δημιουργούνται εμπόδια στις εξαγωγές. Γιατί οι διαπραγματεύσεις είναι χρονοβόρες, γίνονται ανά προϊόν και ανά χώρα και σε ένα χρόνο είναι αδύνατον να επιταχύνουμε την κατάσταση. Θα ήθελα να να πω ότι πέρυσι αυτό το πίνακα ήθελα να σας δείξω τον βρήκαμε τελικά, που δείχνει τους όγκους εξαγωγών προς τη Ρωσία για το 2014 και τη σύγκριση με το 2015 και αυτή είναι η πρόβλεψη των τιμών που βλέπετε. Είναι σκανδαλώδης η, πτώση των τιμών πέρυσι, ιδιαίτερα για τα τρία προϊόντα, δαμάσκηνα, ροδάκινα και νεκταρίνια. Και το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και οι Γάλλοι και οι Ιταλοί συνάδελφοι. η εφαρμογή στις τρίτες χώρες της αντίστροφης στρατηγικής. Ε, αυτό θα πρέπει να ε, προσέξουμε. Επίσης, για μας ήταν πολύ σημαντικό, ένα πολύ σημαντικό ορόσημο, η εφαρμογή των αποσύρσεων των φρούτων για την παραγωγή χυμού. Συγγνώμη, δώστε μου ακόμη μισό λεπτάκι κύριε Πρόεδρε, γιατί είχαμε προβλήματα και με τη διαφάνεια. Δεν πρόλαβα να τα καλύψω όλα. Τι έλεγα λοιπόν. Το ορόσημο για μας ε, ήταν το γεγονός ότι γίνονται αποσύρσεις και χρησιμοποιούνται τα πλεονάσματα για να, παράγουμε χυμό. Αυτό ήταν πολύ χρήσιμο χυμός που διανέμεται σε απόρους, σε φιλαθροπικές οργανώσεις. Η χρήση αυτή ήταν δυνατή, η χρήση λέει δηλαδή, των για την παραγωγή χυμών, κατέστη δυνατή γιατί οι φιλανθρωπικές οργανώσεις δεν χρειάζεται να απορροφήσουν ε, τόσο ρολόσιμα προϊόντα όπως είναι τα πυρηνόκαρπα και καταφέραμε από το καλοκαίρι μέχρι το, τα Χριστούγεννα του 2014 να μετατρέψουμε τα ροδάκινα σε χυμό. Ο χυμός ε, κρατάει πολύ περισσότερο. Θα πρέπει όμως, αν μη τι άλλο, να αποζημιωθούν ε, για το κόστος παραγωγής ε, οι γεωργοί. Επίσης θα πρέπει σεσμικά να προωθούνται τα φρούτα και τα λαχανικά. Θα πρέπει να τονίσουμε τις ευεργετικές ε, συνέπειες που έχουν ε, τα φρούτα και τα σημαντικά ε, περιβαλλοντικά τους αποτελέσματα. Γιατί στην Νότια Ευρώπη έχουμε μεγάλη ανοβρία και ξηρό κλίμα. Είναι σημαντικό λοιπόν να λυθεί και ο περιβαλλοντικός παράγοντας όλα αυτά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ήταν πολύ χρήσιμο που ακούσαμε τις πληροφορίες αυτές απευθείας από το στόμα των παραγωγών. Έχουμε δέκα ομιλητές που ζήτησαν το λόγο. Επειδή έχουμε πίεση χρόνου, ένα λεπτό καθένας. Ο κύριος Γλέζος, παρακαλώ, ένα λεπτό καθένας, δεν έχουμε χρόνο. Το εμπάρκο της ε, Ρωσίας ήταν αποτέλεσμα του εμπάργου που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση πρώτα. Και έχει σημασία ποιος πρώτος ήρξα το χειρών αδίκων. Δεν δικαιολογώ την Ρωσία ύστερα από τη στάση της, αλλά η πολιτική αυτή που δημιουργήθηκε απέναντι στο σύνολο στη χώρα μας είναι τρομερή. Ούτε κονσέρβες έγιναν τα αγροτικά προϊόντα που δεν πουλήθηκαν στην Ρωσία ούτε χυμός έγιναν ούτε γλυκά έγιναν. Μπορούσαν να γίνουν όλα αυτά αλλά ούτε και η αποζημίωση υπήρξε ικανοποιητική. Άρα υπάρχει ένα πρόβλημα που ευθύνεται πρώτα απ' όλα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν από 30 χρόνια ήμουνα εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διαπίστωσα μια πολιτική απέναντι στην Ελλάδα τρομερή οτιδήποτε αγροτικό προϊόν απορρίπτονταν και ρώτησα τους συναδέλφους τελικά τι τη θέλετε την Ελλάδα μου λένε ήλιος, ε, θάλασσα, θάλασσα, φως ναι όλα σύμφωνα δηλαδή μας θέλετε ένα ξενοδοχείο ένα ξενοδοχείο θέλετε την Ελλάδα ξεκάθαρη θέση η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στην Ελλάδα το Αλλά και αυτό είναι σημαντικό. Ο κύριος Φεράν. Merci. Πολύ ενδιαφέρον το θέμα αυτό και ένα θέμα στο οποίο επαναρχόμεθα συνεχώς. Μετά από ένα χρόνο εμπάργο, τα προβλήματα και οι αδυναμίες ε, δυστυχώς ε, καθίστανται ακόμα περισσότερο ανησυχητικές. Και όχι μόνο για τα οποροκυπευτικά. Η διατήρηση του εμπάργου συνεχίζει να επιβαρύνει τους παραγωγούς οποροκυπευτικών αλλά και στα γαλακτοκομικά και στο βόλιο και στο χείριο κρέας. Λοιπόν, ε, τα θέματα τα οποία τίθενται, τίθενται με κατεπήγοντα τρόπο. Κύριε Πρόεδρε, Μπορεί να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν η Ρωσία έχει ενημερώσει τις προϋποθέσεις τις οποίες θα μπορούσε να δεχθεί για να ακυρωθεί αυτό το εμπάργο. Δεύτερον, το Συμβούλιο σκοπεύει να αναδιαρθρώσει τους μηχανισμούς κρίσης για καλύτερη προστασία των παραγωγών έτσι ώστε ε, να υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις ε, και να μην είναι αναγκασμένοι να ξεπουλούν τα προϊόντα τους ε, με τιμές κάτω του κόστους παραγωγής. Ευχαριστώ Ευχαριστώ Πρόεδρε. Στην παρουσίασή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας μίλησε πάρα πολύ για τα μήλα. Τα μήλα είναι εύκολο να αποθηκευθούν γιατί διατηρούνται πολύ καλά σε αλυσίδα κρύου ε, το θέμα είναι τι γίνεται με τα καλοκαιρινά προϊόντα τα οποία δεν μπορούν να διατηρηθούν μακροπρόθεσμα. Ε, Βερίκο, καροδάκινα, ε, κεράσια, δαμάσκινα. Λοιπόν, τι εργασίες έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διευκολύνει τους παραγωγούς των θερινών οποροκυπευτικών. Ο κύριος Νέκοφ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για να επωφεληθούμε και να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τον καλύτερο τρόπο το χρόνο που μου δόθηκε, θα ήθελα να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δείξει πολύ θετική στάση. Αλλά την άλλη φορά, όταν θα είμαι αντιμέτωπο με ενώσει παραγωγών, θα ήθελα να σα πω ότι θα δυσκολευτώ ιδιαίτερω να, πουλήσω, να πουλήσω αυτή τη θετική στάση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η δική μου η χώρα, η Βουλγαρία, μπόρεσε να απολύσει τα προϊόντα της, ε, την περσινή χρονιά πριν το εμπάργκο του Αυγούστου και στη συνέχεια οι επιδοτήσεις δόθηκαν ε, στους πρώτους που τις ζήτησαν. Οι πιο πολλοί παραγωγοί δεν επωφελήθηκαν ύστερα για τις ε, ποσοστώσεις και το γάλα. Δεν υπάρχουν πλέον και πάλι τα αντισταθμιστικά μέτρα τα οποία προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ωφέλησαν πολλούς στη Βουλγαρία. Άρα, να ρωτήσω, ε, έχετε υπόψη σας νέα μέτρα για τους γαλακτοπαραγωγούς ή θα τους αφήσετε και πάλι μόνους τους. Ύστερα, σε ό,τι αφορά την πράσινη εβδομάδα στο Βερολίνο, έγιναν συζητήσεις μεταξύ της ΣΑΝΚΟ και της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Για να μπορέσουν να επιληθούν κάποια προβλήματα, κάποια στοιχεία σε σχέση με την απόρριση. Κυρία Μίλλερ. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έκθεση για τα απορροκυπευτικά. Πιστεύω ότι σε κάποιες περιοχές έγιναν μεγάλες αλλαγές σε ό,τι αφορά την αγορά και σε κάποιες περιοχές ήταν δραματικές και οι αλλαγές των τιμών. Χαίρομαι που η Βραζιλία και η ΙΠΑ ΕΕ, εισήγαγαν πιο πολλά προϊόντα, κοιτώντα τα αριθμητικά στοιχεία. Το θέμα βέβαια τίθεται και σε τι τιμή. Οι διακυμάνσει τη ισοτιμία, οι οποίε ζήσαμε σε σχέση με το δολάριο και το ευρώ, είχαν θετικέ επιδράσει και καταφέραμε κάπω να αντισταθμίσουμε την κατάσταση. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά τα γαλακτοκομικά, το χειρίο και το βόλιο κρέας, δεν είχαμε εκθέσεις. Θα μας κάνετε κάποια σχετική παρουσίαση. Άλλη ερώτηση. Το πρόγραμμα για τα φρούτα στα σχολεία είχε πραγματικά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τις ποσότητες που διοχετεύονται στα σχολεία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ντόρφμαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έκθεση αυτή, αλλά νομίζω ότι κάπως πολύ ρόδινα μας θα παρουσιάζει τα πράγματα σε ό,τι αφορά και τα φρούτα με πυρήνα, το είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι πολλοί παραγωγοί σε τελική ανάλυση θα δουν ένα μεγάλο μηδενικό στα βιβλία τους. Η κατάσταση με τη Ρωσία είναι αυτή που είναι. Όπως είπατε είναι και αισθαντική ισοτιμία με το δολάριο. Αλλά έχουμε και μεγάλες ε, αγορές της ΕΙΠΑ όπου υπάρχουν μεγάλοι προορισμοί εμπορικοί. Γίνεται λοιπόν τίποτα από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να μπορέσει να εξασφαλίσει πιο ευνοϊκή πρόσβαση στην Αμερικανική αγορά. Νομίζω ότι αυτό ήταν η μοναδική λογική προσέγγιση στην παρουσιαφάση αυτή. Ευχαριστώ και ήσασταν και μέσα στο χρόνο σας. Και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα γι' αυτό. Κύριος Μπούντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που υιοθετούμε τέτοια προσέγγιση. Πολύ ωραία λόγια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά τελείως διαφορετικά είναι αυτά που ακούμε από τους παραγωγούς μας. Και κατά το λέω πολύ διαφορετικά. Πού βρήκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη ρόδινη κατάσταση που μας παρουσιάζει, γιατί οι Γεωργοί έχουν πολύ σημαντικά προβλήματα. Παρακαλώ λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κοιτάξει και άλλες αγορές που πλήττονται από το ρωσικό εμπάργκο. Στη Ρουμανία, για παράδειγμα, τα, ο τομέα των παροκυπευτικών έχει κατακλειστεί από προϊόντα τρίτων χωρών. Από χώρες δηλαδή που λαμβάνουν επιδοτήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα προϊόντα του και πολλέ ευθυνέ τιμέ στα μήλα του στη Ρουμανία. Ενώ τα ρουμανικά μήλα μένουν απόλυτα, γιατί δεν έχουν διέξοδο και δεν μπορούν να βρουν αγορά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αναζητήσει νέε αγορές. Είναι η μοναδική εναλλακτική που έχουμε, γιατί σίγουρα το ρωσικό εμβάργο δεν θα καταργηθεί σχετικά σύντομα. Σα ευχαριστώ. Ο κύριο Όγκου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας επισήσω την προσοχή στο εξή. Το ρωσικό εμπάργο επιτάσσει στην Ουγγαρία, Ρουμανία, Σλοβακία, Κροατία, Τσεχία να λάβουν περαιτέρω αποζημιώσεις, το οποίο δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα δυστυχώς. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πότε θα ήταν δυνατή η παροχή των αποζημιώσεων αυτών. Ευχαριστώ. Ε, κύριε κυρία Πετήρ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω παρόμοια ερώτηση με τον κύριο Έρντοσα. Γιατί οι Κροάτες ε, παραγωγοί ε, δεν βρέθηκαν στο κατάλογο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν δικαιούνται αποζημίωση. Και η παραγωγή μανταρινιών, ε, γάλακτος ε, και μήλων έχουν πληγεί ιδιαίτερως. Πώς πρόκειται φέτος να τους αποζημιώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί δεν είχαμε καμία αλλαγή σε σχέση με το ρωσικό εμπάργο. Οπότε η παραγωγή μήλων γάλακτος και νεκταρινιών θα αντιμετωπίσουν προβλήματα αν δεν λάβουν αποζημιώσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, ε, Ευχαριστώ. Έχω μια κάποια σύγχυση για το ποιος ενδιαφέρεται στη Ρωσία σε σχέση με τις κυρώσεις που τους επιβάλλουμε. Οι ηγέτες σε καμία περίπτωση. Δεν τους εκτιμώ ιδιαίτερα, αλλά δεν νομίζω ότι σκοτίστηκε ο Πούτιν για το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόβλημα είναι ότι οι μοναδικοί άνθρωποι οι οποίοι υποφέρουν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν περιορισμένες δυνατότητες και στην Ιρλανδία έχουμε χάσει 230 εκατομμύρια σε επίπεδο εμπορικών συναλλαγών. Σκοτίστηκα για τον κύριο Πούτιν, αλλά αναρωτιέμαι τι νόημα έχουν οι κυρώσεις αυτές και γιατί όχι και εναντίον της Ρωσίας, της Κίνας, της Σαουδικής Αραβίας. Δεν είμαστε ιδιαίτερα συνεκτικοί στη δράση μας. Τέτοιου είδους μέτρα νομίζω ότι βλάπτουν μόνο τους ασθενείς οικονομικά. Ας σταματήσουμε λοιπόν να παίζουμε για πολιτικούς λόγους παιχνίδια με τη ζωή των ανθρώπων. Κυρία Σάνορα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα για μία ακόμη φορά να πω ότι το παράδειγμα της Μούρθια είναι ένα μόνο μικρό τμήμα των προβλημάτων ε, που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί μας. Έχουμε πρόβλημα και με το γάλα, με το βόλιο κρέας, ακριβώς επειδή έχουμε μια κοινή γεωργική πολιτική που προσανατολίζεται αποκλειστικά και μόνο σε εξαγωγές. Θα πρέπει να θεσπίσουμε μέτρα για να αντιμετωπίσουμε έστω και προσωρινά αυτή την κατάσταση που αντιμετωπίζουν χιλιάδες αγρότες μας αλλά στρέφομαι και προς τις, στα μεγάλα πολιτικά κόμματα, στις μεγάλες πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους καλώ να ξεκινήσουμε εκτενή συζήτηση για μια νέα κοινή πολιτική που θα δίνει προτεραιότητα στην εσωτερική αγορά και θα βάλει στο επίκεντρο τα προϊόντα και τα, τις ενισχύσεις σας στους ε, γεωργούς. Και αν διαλέξουμε μεταξύ των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών και της μετανάστευσης, εγώ βλέπω ότι όσο προχωρούν οι συζητήσεις για τις συμφωνίες ε, ελεύθερων συναλλαγών, τόσο περισσότερο αυξάνεται η μετανάστευση και τα χάσματα μεταξύ των δικών μας αγορών και των αγορών των χωρών με τις οποίες έχουμε συναλλαγές. Ευχαριστώ. Εξαντλήσαμε τον κατάλογο των ομιλητών. Οπότε θα ξαναδώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να απαντήσει στις ερωτήσεις και τις απορίες των συναδέλφων. Και για μερικές θα μπορούσατε κάλλιστα να μας στείλετε και γραπτές απαντήσεις, γιατί φαντάζομαι ε, για διεξοδικές απαντήσεις ε, δεν θα είστε προετοιμασμένος, οπότε ό,τι δεν καλύψετε προφορικά, παρακαλώ πιο διεξοδικά γραπτά. Έχετε το λόγο. Thank you, Chairman. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος σε ό,τι αφορά το... την παρουσίαση αυτή την προφορική. Γιατί ξέρω ότι δεν έχετε χρόνο. Να αναφέρω ότι είχαμε μια κρίση πέρσι το, το καλοκαίρι. Χρησιμοποίησαμε το Toolbox σύμφωνα με το άρθρο 119 σε ό,τι αφορά τα μέτρα κατεπήγοντος χαρακτήρα και με τέσσερις ε, πράξεις κατεξουσιοδότηση θέσαμε μέτρα σε εφαρμογή και κάναμε ό,τι μπορούσαμε υπό τις ε, συγκεκριμένες συνθήκες, θεωρώ. Τα αποτελέσματα τα οποία παρατηρούμε τώρα δεν είναι 100% ικανοποιητικά για όλους τους κλάδους, γιατί μιλάμε για αγκούρια, κεράσια, ε, ροδάκινα και μήλα. Βλέπουμε ποιες ε, δυσκολίες υπάρχουν για τις διάφορες ομάδες παραγωγής στο πλαίσιο αυτό. Για το πώς μπορούν όλοι να ικανοποιηθούν παρά το γεγονός αυτό, θεωρούμε ότι οι αγορές στην παρούσα φάση δεν είναι σε μια κατάσταση κρίσης. Ένα δεύτερο στοιχείο εσωτερικά μειώνεται η παραγωγή και στην Ευρώπη. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε αυτή τη μείωση παραγωγής και συγγνώμη, κατανάλωσης απορροκυπευτικών. Γιατί αναφέρθηκε πόσο σημαντική είναι η εσωτερική αγορά, η ενιαία αγορά για τους παραγωγούς. Ένα τρίτο στοιχείο. Το θέμα των τρίτων χωρών. Είναι σημαντικές οι τρεις χώρες ως ε, ενδεχόμενες αγορές εξαγωγής και για αυτές ε, τις χώρες μέλη που είχαν εστιαστεί ως τώρα υπερβολικά στην ε, Ρωσία και στη ρωσική αγορά. Η ρωσική αγορά πάντα ήταν δύσκολη αγορά. Δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζουμε δυσκολίες με μέτρα τα οποία έχει επιβάλει η ρωσική λαμπρά στις εξαγωγές. Άρα, σκοπός μας είναι να υπάρξει διαφοροποίηση σε άλλες θετές χώρες τις πιο πολιτισμένες εξ αυτών κυρίως. Θα ήθελα να πω επίσης ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε και τα προγράμματα προώθησης τα οποία καταστρώνουμε για να δοθεί κίνητρο για τις τρεις χώρες. Εδώ θεωρώ ότι είναι πολύ δυναμικό το πακέτο για την βοήθεια των παραγωγών μας. Όχι μόνο στον τομέα των απορροκυπευτικών, αλλά και στους υπόλοιπους κλάδους. Προκειμένου να εξευρεθούν εναλλακτικέ αγορές και αναπτυσσόμενες ε, αγορές. Και κατά τέταρτον, υπάρχει και το θέμα της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων γενικών διευθύνσεων Σάντε, Grade και Agri, μέσω της πρωτοβουλίας πρόσβασης στις αγορές προκειμένου να αναπτύξουμε συγκεκριμένα μέτρα όπως είναι το SPS που ε, αποκλείουν κάποιους προορισμούς. Αυτό είναι το πακέτο το οποίο είμαστε σε θέση να προσφέρουμε σήμερα και είμαστε φυσικά πρόθυμοι να εμβαθύνουμε στις συζητήσεις και με την Επιτροπή σας και σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Και παρακαλώ να παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς ε, τις αγορές που έχουν πληγεί και επηρεαστεί από το εμπάργκο το ρωσικό και σίγουρα πριν τις θερινές διακοπές θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό. Ε, μας ανησυχεί η πολύ χαμηλή κατανάλωση των φρούτων και λαχανικών ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να βρούμε τρόπους για να τονώσουμε την ε, εσωτερική αγορά αφενός και την εσωτερική κατανάλωση και ταυτόχρονα να συνεχίσουμε την αναζήτηση ε, αγορών και διεξόδων για τις εξαγωγές μας. Επίσης, τον Αύγουστο μας υποσχεθήκατε κάποιες αλλαγές. Αλλά δεν ξέρουμε τι αλλαγές είναι αυτές, ε, γιατί σίγουρα κατάργηση του εμπάργου δεν πρόκειται να λάβει χώρα τόσο σύντομα. Εν πάση περιπτώσει, υποσχεθήκατε ότι θα μα στείλετε γραπτό πιο διεξοδικέ απαντήσει. Θα επανέλθουμε σίγουρα στο σημείο αυτό. Παρακαλώ να παρακολουθούμε ε, τι αγορέ για να δούμε τι τάσει διαμορφώνονται. Αυτά κυρίε και κύριοι. Ολοκληρώνεται η δημόσια συνεδρία τη Επιτροπή. Ραντεβού το απόγευμα στι 3. Προ το παρόν συνεδρία των συντονιστών. Οπότε μία σύντομη ε, διακοπή τεχνική για να περάσουμε στην κεκλεισμένο των θυρών συνεδρίες των συντονιστών. Η δημόσια συνεδρία θα συνεχιστεί το απόγευμα στις 3 στην ίδια αίθουσα. Καλώς μεσημέρι.